ακολουθήσει η ψηφοφορία στο τέλος. Λοιπόν, θα συζητήσουμε κατόπιν το επόμενο θέμα της εκτελέσεις στη Λιβύη. Δίνω τον λόγο στον κύριο Τάνο και ένα λεπτό. Εγώ ποτέ δεν ήμουν απόλυτος ό,τι αφορά τη θανατική τιμή, αλλά μόνο θα πρέπει να ε, καταδικάζονται σε αυτή ε, στιγμή εγκληματίε, όταν ε, έχουν υποστεί δίκαιη δίκη. Αλλά όμω δεν έχω εμπιστοσύνη στο λιβικό δικαστικό σύστημα έτσι όπως έχει σήμερα υπό το δικτατορικό καθεστώς του Γκαντάφη. Είναι εντελώς απαράδεκτο, δεν επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και νομίζω ότι αγνοεί εντελώς τι επιταγέ του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ε, το διακύπημα βέβαια είναι η ε, πετρελαϊκή πόρη της Λιβύης. Ελπίζω ότι η Κομισιόν ε, με κάθε ευκαιρία θα εκφράζει τις ανησυχίες που έχει αυτός ο οίκος για τα, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις ελευθερίες στη Λιβύη. Ε, ξέρουμε τι συνέβη με τις Βουλγάρες νοσοκόμες, ε, οι οποίες καταδικάστηκαν σε θάνατο πριν τελικά απελευθερωθούν μετά από πολλές εκκλήσεις και από εμά και από τη γυναίκα του Γάλλου Προέδρου. Ε, θα πρέπει να προστατεύουμε ε, με κάθε τρόπο την ζωή των Ευρωπαίων πολιτών οποτεδήποτε βρεθούν ε, σε τέτοιες, ε, σε τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Τάνοκ. Ο κύριος Ρωμέβα ή Ρουέδα. Θα χαιρετίζουμε αυτό το ψήφισμα που αφορά τις 18 εκτελέσεις που έχουν λάβει τελευταία στη χώρα στη Λιβύη και τις καταδικάζει. Ε, στη Λιβύη είχαν ξεκινήσει, ξεκινήσει η διαδικασία προς ένα μορατόριο. Πρέπει να ζητήσουμε να συνεχιστεί και να ζητήσουμε διαφάνεια και στατιστικές, γιατί τα πραγματικά νούμερα δεν είναι γνωστά. Ανάμεσα στους 18 αυτούς που θανατώθηκαν υπάρχουν και ε, αλλοδαποί. Θα πρέπει να χαιρετήσουμε αυτό το ψήφισμα που θέτει το θέμα των ε, προσφύγων. Ε, είναι αρμοδιότητά μας ε, και ευθύνη μας ε, και στο πλαίσιο της ε, πολιτικής, μεταναστευτικής μας πολιτικής. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας δεδομένου ότι η Λιβύη δεν έχει υπογράψει συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Η, αναφορά στην αρχή της επαναπρόθεσης και στις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στα δικαιώματα τα άρθρα 18 και 19, είναι απολύτως απαραίτητες. Να προσθέσω και το εξή. Η ιδέα του να χρησιμοποιήσουμε τις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πλαίσιο με την ε, Λιβύη ε, και θα μπορούσε να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε την ε, υπογραφή εκ μέρους της Λιβύης της ε, συνδίκης της Γενέβης και της συνδίκης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το άρθρο 218 της συνθήκη ε, δίνει τη δυνατότητα συμπλήψη τέτοιων όρων σε αυτές τις συμφωνίες και το Κοινοβούλιο θα είναι αυστηρό σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα Ιρουέδα. Η κυρία Βερζιά για δύο λεπτά. Ζητώ συγγνώμη για προηγουμένω, Πρόεδρε. Είχα πραγματικά την εντύπωση ότι δικαίωμαι να μιλήσω για δύο λεφτά. Ε, μαζί με τη Λιβύη υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο ε, συμφωνία, Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα, έτσι ονομάζεται, για την περίοδο 2011-2013, με 60 εκατομμύρια ευρώ για ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, τη υγεία, καθώ και για μια κοινή δράση ε, για την καταπολέμηση τη ε, λάθρομετανάστευση με βάση το κείμενο που έχει μοιραστεί στους δημοσιογράφους. Αυτό το πρωτόκολλο συμφωνίας υπογράφτηκε ε, το Μάρτιο στα πλαίσια του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη στο πλαίσιο του οποίου ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ, ε, συγχωρήστε με, αλλά γελιοποιείται απέναντι στον διεθνή τύπο, ευρωπαϊκό τύπο και αφρικανικό τύπο. Ξέρουμε ότι η Λιβύη είναι κεντρικό άξονα ε, για την μετάβαση μεταναστών προ την Ευρώπη, ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη μιζέρια και να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι φυλακίζονται, εκτελούνται, ε, βασανίζονται. Ε, οι περισσότεροι εγκαταλείπονται στα, στο κέντρο της ρήμου της Αχαράς, χωρίς φαγητό και πεθαίνουν από πείνα και από δίψα. απαντώντας σε μια ερώτηση του, ενός συναδέλφου μου την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος έθεσε αυτό το ερώτημα, απαντάω ότι θα πήγαινε επί τόπου με τον ομόλογο ε, υπουργό της Λιβύης για να δει τι συμβαίνει στη Λιβύη. Αυτό είναι παράδεκτο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και ο Σκαντάφη ε, εμπέζει τις δυτικές δημοκρατίες και οι Ελβετοί φίλοι μας το πλήρωσαν πολύ ακριβά. Η τελευταία πρόκληση είναι το κλείσιμο του γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστίας Προφύγων, την παραμονή των διαπραγματεύσεων. Ε, μας εμπέζουν οι Λίβοι και πρόσφατα συνέβη το ίδιο στα Ιταλικά εδαφικά ε, ύδατα. Μέχρι πού θα πάμε κύριε Πρόεδρε στι διαπραγματεύσει με τη Λιβύη. Ο κ. Μπαρό μα είπε ότι καμία συμφωνία για τη μετανάστευση δεν θα ε, συναφεί στον βαθμό που η Λιβύη δεν έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση τη Γενέβη. Ε, κύριε Επίτροπε, μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει ακριβώς με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ, κύριε Αβερζία. Για ένα λεπτό, κύριο Κάστλερ. Ευχαριστώ. Το 2007 και το 2008 η Λιβύη καταψήφισε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αφορούσε μορατόριουμ στις εκτελέσεις και δεν έδωσε καμία απάντηση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό το ότι τώρα επισήμως αναφέρεται ποια άτομα εκτελέστηκαν. Οποιαδήποτε εκτέλεση είναι μια εκτέλεση παραπάνω από όσε πρέπει. Πρέπει να καταργηθεί η ανθρώπινη φυνή. Είναι απάνθρωπη. Γι' αυτό ζητάμε στο ψήφισμά μας ξεκάθαρα να αλλάξει η κατάσταση, να το πούμε αυτό ανοιχτά και να εργαστούμε από κοινού για να υπάρξει μια αλλαγή εδώ πέρα, να μην έχουμε πλέον μαύρα νούμερα, αλλά ανοιχτά στοιχεία. Τι συμβαίνει και αξιοπρεπείς ποινές για αυτούς που έχουν κάνει κάτι, αλλά όχι υπερβολική τιμωρία ανθρώπων οι οποίοι επικρίνουν το καθεστώς της Τρυπόλεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάσλερ. Τελευταία των συντακτών η κυρία Σάκε. Δύο λεπτά. Εμείς είμαστε μια κοινότητα αξιών ε, και απαγορεύουμε τη θανατική ποινή. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Η Λιβύη όχι μόνο δεν θέλει να καταργήσει θανατική ποινή, αλλά εκτελεί αδιακρίτω. Όπω συνέβη πρόσφατα στι 30 Μαου, όπου 18 άνθρωποι διαφόρων εθνικότητων εκτελέστηκαν με βάση τι ειδήσει που λάβαμε ε, από μια εφημερίδα που πρόσκειται στην ε, κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι παρόλα αυτά η πηγή αυτή είναι αξιόπιστη η πιο σοβαρή τιμωρία, η θανατική ποινή, δεν ε, χρησιμοποιείται μόνο για σοβαρά εγκλήματα. Απαγορεύεται και η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεστη και αυτές, αυτές οι δράσεις οδηγούν σε θανατική ποινή. Νομίζουμε ότι η Ελληνική πρέπει να ενταχθεί στη διεθνή κοινότητα και να βγει από την απομόνωση, να βγει και ο λαός από την απομόνωση στα χέρια αυτού του αυτο, αυταρχικού καθεστώτος. Εμείς το 2003 ε, ήραμε τις... Ε, κυρώσει εναντίον της χώρα και ξεκινήσαμε το 2007 τι διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, συζήτηση με τη Λιβύη. Αυτό είναι δυνατόν μόνο στο βαθμό που η Λιβύη ε, σεβαστεί τις ε, βασικές ελευθερίε και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων της. Το κλείσιμο του γραφείου της ΥΠΑ στην Τρίπολη είναι ένα, μια επιπλέον χειρονομία της Λιβύης που την αποσπά από τους κόλπους της διεθνούς κοινότητας δεδομένων των συνεχών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να έχει η έδρα στο Συμβούλιο ασφαλεία του ΟΗΕ. Θα πρέπει ε, μόνο τα κράτη που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα να έχουν έδρα. Αλλιώς όλος ο φορέας, όλο το σώμα αυτό χάνει την αξιοπιστία του. Όπως παραδείγματο χάρη όταν το Ιράν ήταν μέλος ε, του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων των Γυναικών του ΟΗΕ, κάτι που πραγματικά σπηλώνει την αξιοπιστία και το κύρος της οργάνωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει έκκληση στη Λιβύη να καταργήσει την, την θενατική ποινή και να σεβαστεί τα διεθνή πρότυπα. Και όλα τα κράτη-μέλη όταν εκδίδουν ε, υπηκόους προς τη Λιβύη θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι ευθύνες τους, γιατί πολύ πιθανό οι άνθρωποι αυτοί να πέσουν θύματα απάνθρωπης μεταχείρισης. Ευχαριστούμε κυρία Σάκη. Ακολουθούν οι ομιλητές των ομάδων. Η κυρία Μακοβέη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ λυπούμε για την εκτέλεση 18 τόμων στην Λιβύη το Μάιο του 2010 και ζητώ την κατάργηση θανατικής ποινής. Η Λιβύη χρησιμοποιεί θανατική ποινή για να περιορίσει την ελευθερία του λόγου και του συνέρχεστε στη χώρα και δεν μπορούμε να καταγράψουμε τις περιπτώσεις. Όμως η Human Rights Watch πήρε συνέντευξη με έναν κρατούμενο και είπε πως τελευταία στιγμή μετετράπη η ποινή του σε ισόβια. Σύμφωνα με τον Αλ Σαρίφ, το Λαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε αυτόν και δύο άλλους για οργάνωση πολιτικής ομάδας που ήταν κατά της επανάστασης της Αλφατάχ. Το Ανώτατο Δικαστήριο Εβεβαίωσε αυτές τις ε, ποινές, αλλά τελευταία στιγμή, το Φεβρουάριο του 2002, αφού είχαν περάσει μία ώρα με δεμένα τα μάτια δεμένοι σε έναν πάσαλο, η ποινή τους μετατράπηκε, σύμφωνα με την Αλσαρίφ. Από όσα ακούγονται, πάνω από 200 άνθρωποι αυτή τη στιγμή αναμένουν εκτέλεση Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει να διάλογο για αυτά τα θέματα με την Λιβύη. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Η κυρία Κρατού για ένα λεπτό. Η θανατική ποινή είναι η πιο απάνθρωπη και βάρβαρη κύρωση η Λιβύα είναι μία από τις 12 χώρες ε, που χρησιμοποιούν ακόμα τη θανατική ποινή, παρόλο που αυτό δεν εγκρίνεται ούτε από τον ΟΗΕ, ούτε από την πλειοψηφία των κρατών του κόσμου. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσει ακόμα περισσότερο για την κατάρριξη της θανατικής ποινή και ταυτόχρονα έχει το καθήκον να αυξήσει τις πιέσεις ε, επί της Λιβύης προκειμένου να καταργηθεί η θανατική ποινή, όχι απλώς να μην χρησιμοποιείται. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά, ιδιαίτερα στα δικαιώματα των αλλαδαπών πολιτών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν δικαίωμα ούτε σε διερμηνέα, ούτε σε μετάφραση των ε, δικογράφων. Ε, δεν, έρχονται σε, δεν τους δίνεται δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αντιπροσώπους από τη χώρα τους, με τις οικογένειές τους. Ε, δεν έχουν πρόσβαση σε χρήματα. Ε, δεν ενημερώνεται καν η οικογένεια των θυμάτων πολλές φορές. Η Λιβύη λοιπόν θα πρέπει να σέβεται τους ε, διεθνείς ε, κανόνες περί ισότητας ενώπιον του νόμου κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κρετού να ακολουθούν οι υπόλοιποι ομιλητέ. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Σόνικ για ένα λεπτό. Τέλος Μαΐου ε, εκτελέστηκαν 18 άτομα Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 200 άτομα που βρίσκονται στη φυλακή και ορισμένοι από αυτού περιμένουν να εκτελεστούν ω νούπο. Αυτό ο αριθμό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Ε, η Λιβύη παίζει με διπλά στοιχεία. Άλλα νούμερα μας λέει εμάς, άλλα λέει στον ΟΗΕ και παράλληλα συνεχίζει τις δολοφονίες. στην πραγματικότητα υπάρχει απαγόρευση ε, της χρήσης της θανατικής ε, και μπορεί να χρησιμοποιείται ε, μόνο για πολύ σοβαρά εγκλήματα. Παρ' όλα αυτά η Λιβύη θανατώνει για ναρκωτικά, για, ακόμα και για την, την ελευθερία της έκφρασης. Και αυτό είναι ε, αδίκημα για τη Λιβύη που επισύρει τη θανατική ποινή. Ε, θα θέλαμε ε, να επικυρωθεί από τη Λιβύη η Σύμβαση της Γενέβης, καθώς και άλλες συμβάσεις που προσπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο συν, κύριος Συνδυσίν. Ευχαριστώ. Η προστασία της, της αξιοπρέπειας είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Και όμως στις περισσότερες χώρες, ε, ακριβώς γι' αυτό στις περισσότερες χώρες υπάρχει μορατόριο της θανατικής ποινής. Η χρήση της θανατικής ποινής μας επαναφέρει στο μεσαίωνα. Οι εκτελέσεις είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κλείσιμο του γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστίας και η απέλαση 26 υπαλλήλων από τη Λιβύη ε, είναι μια κατάφορη παραβίαση όλων των διεθνών συμβάσεων. Οποιαδήποτε προϋπόθεση για τη σύναψη συμφωνίας με τη Λιβύη θα πρέπει να είναι η, υπογραφή από τη Λιβύη της ε, σύμβασης ε, και των πρωτοκόλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μας τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδη σημασία και θα πρέπει να τα εγγυάται και η Λιβύη. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Κόρχολα για ένα λεπτό. Κυρία Κόρχολα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ανεπίσημες επαφές με τη Λιβύη και υπάρχει και σύμφωνο φωνία επί μετανάστευσης. Κάτι προβληματικό αυτή τη στιγμή γιατί η Λιβύη δεν έχει λάβει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ε, υπό τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε 18 εκτελέσεις, περίπου 200 άτομα έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Ορισμένοι από αυτούς είναι αλλοδαποί. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Λιβύη θα επικυρώσει τη σύμβαση για τους πρόσφυγες, κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να συντονιστούν με τον ΟΗΕ, να σεβαστούν τις συμβάσεις του ΟΗΕ και να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να επαναπαστρεφιστούν. E, για εμάς τους Ευρωπαίους η θανατική ποινή είναι κάτι το πραγματικά ανήκουστο που δεν διαθέτουμε πλέον στην πολιτική μας Γι' αυτό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Λιβύη είναι ιδιαίτερα απεχθές. Ειδικά όταν αναφέρεται σε αλλοδαπούς που δεν έχουν καμία σχέση με τη Λιβύη. Η τελευταία λοιπόν ενημέρωση για εκτέλεση 18 ατόμων μεταξύ των οποίων και Αιγύπτιοι, Νιγηριανοί και τα είναι πολύ απεχθής ειδικά εφόσον δεν είχαν και κάποια ε, βοήθεια στη διάθεσή τους, ε, προξενική βοήθεια, διερμηνείς, δικηγόρους κτλ. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα την επόμενη εβδομάδα στην αντιπροσωπεία για το Μαγκρέμπ με τους εκπροσώπους από τη Λιβύη και πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέντα, πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο, θα ήθελα να σας πω το εξή προσωπικά. Σχεδόν οι μισοί συνάδελφοι ε, διαβάζουν κείμενα. Και εδώ ανάβει ένα λαμπάκι slow down. Παρακαλώ μην διαβάζετε πιο γρήγορα από όσο σκέφτεστε, γιατί διαβάζετε τότε πιο γρήγορα όσο μπορούν να σκεφτούν οι διερμηνείς. Και ό,τι έχετε γραμμένο μπορείτε να το δίνετε στους διερμηνείς για να τους διευκολύνετε τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσυπογράφει τις απόψεις τις οποίες εξέφρασαν οι συνάδελφοι ε, για τις πρόσφατες εκτελέσεις 18 ατόμων στη Λιβύη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τις εκτελέσεις διότι αυτό δεν συνάδει με τις αξίες μας. Θεωρούμε ότι η θανατική ποινή είναι βάναυση και απάνθρωπη εάν δεν υπάρχουν ε, αποτρεπτικά μέτρα για την κλιματική συμπεριφορά και θεωρούμε επίσης ότι είναι κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερως ενοχλημένη από το γεγονός ότι οι εκτελέσεις έγιναν εβδομάδες μετά από την εκλογή της ε, Λιβύης ε, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. έγινε διάβημα προ τι Λιβικέ αρχές για να εκφράσουμε την καταδίκη των θανατικών ποινών και να υπενθυμίσουμε στη Λιβύη τη νομική της υποχρέωση να προσφέρει όλες τι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίσει μια δίκαιη δίκη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 14 για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα τα οποία επικύρωσε η Λιβύη το 1970. Επίσης, ενθαρρύνουμε τη Λιβύη να ετοιμάσει μορατόριου ώστε να καταργηθεί η θανατική ποινή για οποιαδήποτε, ε, για οποιοδήποτε αδίκημα. Η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με το ε, Λιβύη θα μας αποδώσει τη νομική βάση η οποία είναι απαραίτητη για να έχουμε συνεργασία σε όλα τα θέματα ε, ποινικού δικαίου και οι διαπραγματεύσεις για αυτή τη συμφωνία πλαίσιο προχωρούν καλά. Έγινε ο 7ο γύρο διαπραγματεύσεων την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρίπολη και μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έγινε πολύ σημαντική πρόοδο, κυρίω σε πολιτικά θέματα. Τέλο, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί πλήρω ότι κάποια θέματα είναι πολύ δύσκολα στι σχέσει με τη Λιβύη, Ωστόσο, είμαστε δεσμευμένοι και θέλουμε να ε, προχωρήσει περαιτέρω ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης επί τη βάση αμοιβαία εμπιστοσύνη, για να έχουμε με επικοδομητικό τρόπο αντιμετώπιση όλων των θεμάτων όπως είναι ένα τόσο ευαίσθητο θέμα ε, που έχουμε σε αυτή την περίπτωση. παρά το γεγονό ότι θεωρούμε ότι αυτέ οι σχέσει έχουν κάνει ένα θετικό βήμα προ τα μπρο, θέλουμε να υπάρξουν οι σχέσει αυτέ επί τη βάση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Πέρα στη συζήτηση θα ξεκινήσουμε τώρα την ψηφοφορία. Καταρχά θα ψηφίσουμε τι έξι προτάσει ε, ψηφίσματο για το Κονγκό. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφοφορία για έξι προτάσεις ψηφίσματος για το ΛΕΠΑΛ. Έχουμε